Welcome to Γεια σας, σας καλωσορίζω. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για δύο λόγους. Ακουστικά παρακαλώ, να τα χρησιμοποιήσετε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εγώ είμαι ένας από τους 500, τα 550 εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν Ισπανικά. Άρα θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Το δεύτερο είναι γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα διερμηνέων ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Mi colega η συνάδελφος η Γκεζίνε Μάισνερ μας είπε ότι ο Αλέν Καντέκ δεν πόρεσε να παρευρεθεί εδώ. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να προεδρεύσω σε αυτό το εξαιρετικό πάνελ ομιλητών. Ε, λυπούμεθα που δεν βρίσκεται εδώ ο Αλέν, αλλά θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπροσώπους, τους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους μου, ευρωβουλευτές. Εφόσον άλλαξε λοιπόν η σειρά παρουσίασης, θα μιλήσω και εγώ στην πρώτη φάση συζήτησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τρία τέταρτα του πλανήτη ε, αφορούν το νερό, δηλαδή απαρτίζονται από ύδατα και σε όγκο και σε ε, κυβικά. Πρόκειται για το 70% των υδάτων που απαρτίζουν τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο με 25 χώρες και περιφέρειες, θαλάσσιες περιφέρειες και βεβαίως αυτό περιλαμβάνει και τα Κανάρια νησιά που είναι απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή. Πέρα λοιπόν από την ε, νομιμότητα και τη θεμητότητα συμμετοχής μας θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στον αλληλευτικό τομέα τι εννοούμε όταν μιλάμε για διαχείριση των ωκεανών, διακυβέρνηση των ωκεανών, τι σημαίνει αυτό, τι προϋποθέτει. Θα ήθελα να σας μιλήσω, να σας σκιαγραφίσω τι σημαίνει καλή διακυβέρνηση των ωκεανών. Η καλή διαχείριση περιλαμβάνει και αφορά την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αλία δεν έχει σύνορα και αυτό ακριβώς σημαίνει και γι' αυτό υπάρχει κοινή αλλιευτική πολιτική. Άρα η διασυνοριακή διάσταση των ωκεανών δείχνει ότι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα, στο πιο ευρύ πλαίσιο αλλά και πιο περιορισμένο. Καλή διαχείριση επίσης σημαίνει σωστή συμμετοχή των οικονομικών φορέων. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω ιδιαίτερα. Θα πρέπει να ακούσουμε την επιστημονική κοινότητα της ΜΚΙΟ και ολόκληρο τον τομέα και θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να συμμετέχουν ε, δραστικά γιατί θα δράσουμε όχι για τους οικονομικούς φορείς αλλά με τους οικονομικούς φορείς. Το δεύτερον ε, αφορά την ανάγκη χρήσης εύκολων όρων που να αποτελούν επίκληση. Δηλαδή μιλάμε για εκφόρτωση, για χώρους εκφόρτωσης φόρτωσης και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Δεν πρέπει όμως να εμείνουμε στην ορολογία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα και να μην χρησιμοποιείται η δημαγωγία για το απόλυτο κέρδος, διότι αυτό θα μας πλήξει άμεσα. Οι θαλάσσιες ε, περιφέρειες, θαλάσσιες περιφέρειες, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιφέρειες αποτελούν χήμερα. Έχουν ευεργετήματα βεβαίως και αποτελούν ένα μέσο διαχείρισης αλλιευτικών δραστηριοτήτων και για μία προστασία των θαλάσσιων περιοχών, αλλά δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Πέμπτο σημείο. Δεν θα πρέπει να εντυπωσιάζουμε με όρους οι οποίοι είναι δυσνόητοι και δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Εδώ ε, αναφέρομαι στο MSY, το οποίο για πολύ καιρό απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, τους επιχειρηματίες, τους επιστήμονες και τους οικονομικούς φορείς. Και νομίζω ότι σήμερα καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να δούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε να το αποδώσουμε καλύτερα και να το θέσουμε σε φαρμαγή. Δηλαδή την μέγιστη αυτή βιώσιμη απόδοση. Μη χρησιμοποιώντας μη χρησιμοποιώντας ε, ε, περίεργους όρους. Επίσης υπάρχει ένας ε, άλλος όρος για την βέλτιστη χρήση των ωκεανών. Έχει μεγάλη σημασία η χρήση ε, των πόρων όπως προβάλλουν οι εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς. Μιλώ για τις ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, για την αρχή της βιοπικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη αποφάσεων στο μέα της διαχείρισης της αλίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε και να ενισχύσουμε τα ε, παγκόσμια μέσα που έχουμε ή περιφερειακά μέσα. Γιατί πολύ συχνά όταν οι προσπάθειες δεν αποδίδουν δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομοθεσία αλλά υπάρχει θέμα εφαρμογής του νόμου. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με την αλληλευτική πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχουν ορόσημα και πλαίσια για τον ευρωπαϊκό αλληλευτικό στόλο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία εάν λάβουμε υπόψη τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της βιωσιμότητας ε, χρήσης του ε, στόλου μας, ο οποίος δεν πρέπει να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει η ηγετική θέση έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες και τις προκλήσεις μέσα στα πλαίσια της βιωσιμότητας των πόρων. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την αλία και τον αλλιευτικό στόλο, η υπεραλίευση, οι κλιματικές αλλαγές, καθώς και η παράνομη, αδήλωτη και άναρχη αλίευση. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες προσπαθήσαμε να απαλείψουμε αυτή τη μάστιγα μέσα στα πλαίσια της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τρίτες χώρες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τα αλλιεύματα, τα παράνομα αλλιεύματα να μην φτάνουν σε εμάς. Αυτό αφορά και το ένατο σημείο που είναι και το τελευταίο. Τι γίνεται σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πρόκληση, πρόκληση στον τομέα της ηχθειοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα όταν οι θάλασσές μας πλήττονται από τις θαλάσσιες μεταφορές και την εκμετάλλευση των πρώτων υλών, την μόλυνση των θαλασσών και τις κλιματικές αλλαγές. Για όλους αυτούς τους λόγους που είναι ε, ολίγιστη σε σχέση με το σύνολο, θα πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση των ωκεανών. Η υγεία των ωκεανών έχει μεγάλη σημασία για την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους διαχειριστούμε και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους πόρους, να έχουμε καθαρούς ωκεανούς ε, παραγωγικούς, ασφαλείς και υγιείς και προπαντός προστατευόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και τώρα θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδιοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Ο κάθε ένας από τους ομιλητές θα πρέπει να μιλήσει γύρω στα τέσσερα λεπτά. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην Αιτάρ Ματσάδο που είναι καλός φίλος και Γενικός Διευθυντής στην ε, Γενική Διεύθυνση Αλίας και Θαλασσών. Ευχαριστώ αγαπητέ Γάμπριελ και αξιόλο, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πίτρο Πεβέλα, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι η συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης ε, μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Και σήμερα έχουμε τόσους νέους εδώ είναι επίσης κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας χαροποιεί. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα εδώ στο Κοινοβούλιο είναι προήμιο σύστασης μιας επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Αλία και τους ωκεανούς. Νομίζω πως θα ήταν καλή μια ιδέα για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία και θα μας ωφελούσε όλους. Ευχαριστώ και συγχαίρω πολλούς ε, ευρωβουλευτές για τις προσπάθειες ε, που έχουν κάνει όπως, που έχουν κάνει, όπως η κυρία Ροντούστ και ο κύριος Σάντους για να είναι προτεραιότητα το θέμα αυτό για το Κοινοβούλιο. Όπως είπαν και διάφοροι ομιλητέ ήδη προηγουμένως, οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι ζωτική σημασία για όλους μας. Είτε μένετε κοντά στην παραλία είτε στο εσωτερικό μιας περιοχής είναι ζωτική για την ε, ζωή. Αλλά ε, υφίστανται πιέσεις, είναι ευαίσθητοι και χρειάζονται καλύτερη προστασία, φροντίδα, διαχείριση γιατί τους έχουμε παραμελήσει συνολικά ως παγκόσμια κοινότητα για πολλά χρόνια. Εμείς πριν από τέσσερα χρόνια, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτήσαμε τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους αν θεωρούσαν το διεθνές πλαίσιο για την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών το τρέχον τότε ήταν επαρκές και ε, αποτελεσματικό σχεδόν όλοι απάντησαν όχι. Όχι επειδή το υπάρχον ε, διεθνές πλαίσιο που έχει κέντρο τη Σύμβαση των Ηνωμένων για το δίκαιο των θαλασσών δεν είναι σωστό, αλλά γιατί υπάρχουν κενά από πλευράς διεθνών ε, μέσων, ορισμένα είναι και ανεπαρκή και αναποτελεσματικά και δεν υπάρχει επαρκή συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων που έχουν δημιουργηθεί ε, όλα αυτά τα χρόνια. Και μόνο μέσω ισχυρής διεθνούς συνεργασίας που ε, στη σημερινή συγκυρία δεν είναι από τα πιο δημοφιλή ε, θέματα. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, παγκόσμια φύση των προβλημάτων αυτών. Μόνο ενωμένοι, μόνο συνεργαζόμενοι μεταξύ χωρών, μεταξύ, πέρα από σύνορα μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή για πρώτη φορά η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Βέλα και της ε, υπάτης εκπροσώπου Μογκερίν. Μόνο λοιπόν που τότε, τότε που για πρώτη φορά υπήρξε ένα έγγραφο για την ε, παγκόσμια διαχείριση των ωκεανών υπήρξε μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η ε, κατάσταση όπως ήταν και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, όπως είπε και ο Επίτροπος Βέλλα στην εισαγωγή του, δημοσιεύουμε για πρώτη φορά μια έκθεση προόδου για το σε τι βαθμό και με το τι τρόπο επιτύχαμε τους στόχους που θέσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Στην έκθεση αυτή είναι προσβάσιμη. Θα δείτε ότι οι υποσχέσεις μας μετατρέπονται σε δράση και στον ε, αλληλευτικό τομέα. Λοιπόν, να τονίσω την πολύ σημαντική συμφωνία, καταρχάς, που συνήφθη τον περασμένο Οκτώβριο για μια νέα συμφωνία. Λοιπόν, μια νέα συμφωνία λοιπόν για την αλληλεία στον, στην Αρκτική που απαγορεύει την ε, αλληλεία για 16 χρόνια ε, στην κεντρική Αρκτική και ε, θα μπορούσε κατόπιν να επεκταθεί άλλα 16 χρόνια αυτή η απαγόρευση αν συμφωνήσουν οι συμβαλόμενοι. Δεύτερον, η Ένωση και όπως είπε ήδη ο Γκάμπριελ έχει πολεμήσει σκληρά για να εξαλειφθεί η παράνομη αλληλεία και έχουμε αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό όργανο σε ενωσιακό επίπεδο που μας επέτρεψε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά πολλών ε, από τους εταίρους μας και να εξαλειφθεί η παρουσία αλλιευμάτων που έχουν αλλιευθεί παράνομα στις ευρωπαϊκές αγορές. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε εξάλλου ένα δίκτυο εταιρικών ε, συμφωνιών με τρίτες χώρες για θέματα αλλίας και αυτό βασίζεται στη νέα κοινή ελευτική πολιτική που θέτει στο κέντρο της προσοχής μας την βιωσιμότητα και την ε, υγεία των ε, ε, διαφόρων αλλιευτικών ειδών. Έχουμε συμφωνίες με τη Μαυριτανία, με το Μαρόκο, το Πράσο Κροτήριο, τη Γουνέα Μπισάου και επίσης σε αυτή τη νέα γενιά συμφωνιών υπάρχει και η διάσταση της θαλάσσιας οικονομίας, της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης. Τέταρτον, προωθούμε μαζί με τους εταίρους μας την ανάπτυξη μια βιώσιμη γαλέζια οικονομία. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και ορισμένοι από του ομιλητέ στην ανακτήρια εκδήλωση το ανέφεραν. Πρέπει όμω να είμαστε προσεκτικοί. Η γαλάζια οικονομία πάντα πρέπει να εξετάζεται από την πλευρά της βιωσιμότητας για να αποφύγουμε τα λάθη που έγιναν για την ε, γεωργία και οτροφία. Τώρα, για να είναι αξιόπιστη σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε αξιόπιστες στο εσωτερικό μας. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τις προσπάθειες που έχουμε μαζί με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο και με τον κλάδο της αλίας. Και έχει υπάρξει τρομερή πρόοδος, ούτως ώστε τα θέματα να παραμείνουν σε υγιή κατάσταση. Ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τα αποθέματα σε τόσο βιώσιμο επίπεδο όπως τα έχουμε σήμερα. Με συγχωρείτε, ήδη ξεπέρασα το χρόνο μου. Θα σταματήσω εδώ. Αλλά θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε και περαιτέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω που συνεργανώνετε με την Επιτροπή αυτή την εκδήλωση και με χαρά να συμμετάσχω στην περαιτέρω συζήτηση και σα ευχαριστώ πολύ.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 σπάσουμε τα στεγανά και να δούμε διακλαδικά, διατομεακά το θέμα των ωκεανών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουμε συλλογική ευθύνη να προσφέρουμε λύσεις ε, για ασφαλείς, ε, υγιείς, βιώσιμους στη διαχείρισή του ωκεανού. πώ θα βρούμε καινοτόμου τρόπου να διαχειριστούμε του ωκεανού, εμεί στηρίζουμε τη λεγόμενη διατομιακή προσέγγιση. Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των τομέων. Είναι μια συνεργατική ε, προσέγγιση που τη βλέπουμε και στην έκθεση πρόοδου για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών που εγκρίναμε στις 15 ε, Μαρτίου μετά από δύο χρόνια δράση και μετά το policy paper που είχε κατατεθεί στα τέλη του 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται στην διαχείριση των ωκεανών και στο θαλάσσιο πολυμερέ σύστημα γιατί θέλουμε να εφαρμοστούν σωστά οι φυστάμενοι κανόνε και να πληρωθούν τα διοικητικά κενά. Θέλουμε επίση διευκόλυνση τη συνεργασία ε, και ανάληψη νέων πρωτοβουλειών. Είμαστε πεπισμένοι πως οι ωκεανοί θα πρέπει να είναι υψηλά στο διεθνές θεματολόγιο στο πλαίσιο και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Ε, όταν είναι ρευστά τα πράγματα, και όταν υπάρχει μια παγκόσμια βεβαιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στο να είναι προβλέψιμος, ε, αξιόπιστος πρωταγωνιστής ε, στο διεθνές προσκήνιο, σε στενή συνεργασία βέβαια και με άλλους φορείς. Στηρίζουμε μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες. Και αυτό το δείχνει και η υποστήριξη που παρέχουμε στο θεματολόγιο του 2030 και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και υπάρχει και η παγκόσμια στρατηγική εσωτερικό έγγραφο της Ένωσης για την ε, κοινή εξωτερική πολιτική. Εκεί οι ωκεανοί έχουν μεγάλη προτεραιότητα. Τα δύο τελευταία χρόνια προβάλαμε περισσότερο και το θέμα της ε, παγκόσμιας διαχείρισης των ωκεανών στις ε, συνομιλίε με τρίτε χώρε, στα περιφερειακά μας προγράμματα και στρατηγικές και αυτό το πράξαμε διότι πιστεύουμε πως η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, για ασφαλείς οδούς, ε, εμπορίας αγαθών, για ένα ασφαλές θαλάσσιο περιβάλλον και για τη διαχείριση των ωκεανών συνολικά υπέρ της υγείας και της σταθερότητας ε, συνολικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως μόλις είπε ο καλός μου φίλος ε, Ζωάου, Αγιάρ Μασάδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά πολλές χώρες να καταπολεμήσουν την παράνομη αλία στα εδάφη για να υπάρχει μεγαλύτερη ε, διακυβέρνηση των ωκεανών συνολικά στις θαλάσσιες περιοχές. Επίσης υπάρχει συνεργασία για την περισυλλογή των μικροπλαστικών και των θαλάσσιων απορριμμάτων σε συνεργασία παραδείγματος χάρη με τις ασιατικές χώρες, την Νοτιοανατολική Ασία, με τις χώρες του ΑΖΕΑΝ. Επίσης έχουμε συνεργασία για την προστασία της Αρκτικής και της Ανταρκτικής όπως προαναφέρθηκε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της έρευνας, της συλλογής δεδομένων. Έχουμε επενδύσει σοβαρά στην επιστημονική συνεργασία και στα προγράμματα δορυφορικής παρακολούθησης μέσω του Κοπέρνικους, για παράδειγμα. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε ενεργοί και ε, να αναλαμβάνουμε τον των προτέρων δράση για την προστασία των θαλασσών ε, ε, και προστατεύοντας κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, Ατλαντικό, Ασία. Θέλουμε να Προωθήσουμε επίσης ε, το σεβασμό στα νομικά δεσμαυτικά μέτρα και συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουμε να προωθήσουμε το διάλογο για όλα αυτά τα θέματα. Είναι όλες αυτές πρωτοβουλίες που δείχνουν πώς ανταποκρινόμαστε συνολικά στο θεματολόγιο 2030 και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε και μεταξύ αυτών το στόχο 14 που αφορά τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση ωκεανών, θαλασσών ε, και θαλάσσιων πόρων εν γέννη. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη όμω είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ του και θα πετύχουμε πρόοδο στον στόχο 14 αν έχουμε πρόοδο και στου άλλου παρότι ο 14ος αυτός στόχος έχει πολλά να προσφέρει για την επίτευξη και των άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχει πρόκληση λοιπόν να λάβουμε κατεπίγουσα δράση για να σώσουμε τους ωκεανούς. Πρέπει όμως να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία και ε, να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί. Έχουμε συλλογικέ ευθύνε. Ε, δεν πρέπει να αποστρέφουμε το βλέμμα από αυτές. Επίσης, ζωή στους ωκεανούς, ε, η ζωή των ωκεανών δεν είναι απλά αυτό. Είναι η ζωή του ίδιου του ανθρώπου, είναι η ζωή ε, των τοπικών κοινωνιών που ζουν δίπλα στη θάλασσα, που συμβιούν ε, ουσιαστικά με τους ωκεανούς. Ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ευημερία, συνολικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όλα αυτά θα προστατεύσουν τον πλανήτη μας. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας συνεισφορές και προτάσεις γιατί μπορούμε να πετύχουμε μόνο αν συνεργαστούμε ε, όλες οι κοινωνίες και όλοι οι παγκόσμιοι εταίροι και οργανισμοί. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να μιλήσει για τρία λεπτά το ανώτερο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Χωσέ Ινάσιο Φαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Γκαμπριέλ Μάτο. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχήν τον αγαπημένο μου επίτροπο Καρμένου Βέλα και σας ευχαριστώ για την εργασία σας για την διατήρηση των ωκεανών μας. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω την Γκεζίνε Μάισνερ, τη συνάδελφο και τέλος, για να μην ξεχάσω κανέναν, θα ήθελα να χαιρετήσω τον συνάδελφο Ρικάρδο Σάντος, ε, του τη συνάδελφο Κλάουδια Μοντέρο Γκιάς και τον ε, Ζουάου Μασάδο, ο οποίος ε, ήταν υπεύθυνο για την αλλιευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η Πορτογαλία έχει μακρά παράδοση στους ωκεανούς και έχει πολλούς ανθρώπους στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Κοινωνία των Πολιτών. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται την ευθύνη της για την χρήση των ωκεανών μέσα στα πλαίσια της ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και δυνάμει του στόχου 14. Μετά το τέλος της διαδικασίας διακυβέρνησης το 2017 ανέκυψε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να μιλήσω για τρία στοιχεία άξονες για να παραμείνει ο πλανήτης μας γαλάζιος. Ε, διπλωματία για το κλίμα, προστασία του περιβάλλοντος και μπλε πόροι, οικονομικοί Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την υπερεκμετάλλευση των πόρων για να μην υπάρχει τέτοια πίεση στα λιευτικά αποθέματα. Θα πρέπει να έχουμε πιο συνειδητή αλία που να μην βασίζεται στο κέρδος και την διφαγία αλλά τη βιωσιμότητα. Έτσι μόνο οι ωκεανοί θα παρέχουν πόρους για τους Ευρωπαίους. Και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε και την υδατοκαλλιέργεια. Μία άλλη έννοια είναι οι επιπτώσεις του Brexit για να δούμε τι θα γίνει με την απώλεια υδάτων χωρίς να υπάρξει πίεση ως προς τα αλλιευτικά αποθέματα άλλων περιφερειών. Θα ήθελα να σταθώ στην έρευνα και την ενέργεια, την καθαρή ενέργεια και την βιοτεχνολογία έτσι ώστε η έρευνα να μετατραπεί σε καινοτομία και να δημιουργηθούν και νέες ευκαιρίες στην πλέ οικονομία. Πιστεύω ότι η, ο η ενέργεια των ωκεανών θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτροπή ε, διοξιδίου του άνθρακα και να δημιουργήσει και 500.000 θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να μειωθεί και η χρήση ορυκτών καυσίμων. Όμως ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτή η εκμετάλλευση οδηγεί σε κλιματικές αλλαγές. Οι Ευρωπαίοι τόνισαν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν σε μία οικονομία χαμηλής χρήσης του άνθρακα έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπεράκτιες ε, επιχειρήσεις εξόριξης και να υπάρχει χαμηλή χρήση ή και μηδενική του άνθρακα. Εάν ε, συνεχίσουμε να ρίχνουμε ε, λίματα καθώς και όσο υπάρχουν πετρελαιοκυλίδες ή ε, ρήψη φαρμακευτικών προϊόντων, τότε θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα υγείας. Αυτό αφορά όχι μόνο περιβαλλοντική, αλλά και οικονομική ζημία. Έχουμε έναν νέο κανονισμό για τη χρήση εξοπλισμού μοναδικής χρήσης και θα οδηγήσει σε αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά με βάση αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μόνο το μέλλον θα το ε, δείξει. Αυτό που μετράει τώρα είναι να μαζεύουμε τα λύματα και να τα δεσμεύουμε, τα λύματα που υπάρχουν στους ωκεανούς και να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου, μεθανία και μαύρου άνθρακα. Επίσης, η θαλάσσια δραστηριότητα οδηγεί σε συγκεκριμένες διαρροές, πετρελαιοκυλίδες και ούτω καθεξής. Και αυτό ε, έχει μεγάλη επιρροή και στον ευτροφισμό και στα πλανκτόν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά, αυτά στις αρνητικές απόρριες θα πρέπει να έχουμε αποκλειστικές οικονομικές ε, ζώνες που να είναι 25,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο μέσα στα πλαίσια της ε, φιλόδοξης οικονομικής διακυβέρνησης των ωκεανών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ένας φάρος δράσης στα πλαίσια του Διεθνούς Θαλάσσιου Οργανισμού. Τέλος, ε, για την Αρκτική, οι κλιματικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε ε, αλλαγές μεταξύ Βόρειου Ειρηνικού και Βόρειου Ατλαντικού. Θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε την ε, οικολογική καταστροφή με τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα πυρηνικά πλοία. Έχουμε έναν εξαιρετικό γαλάζιο πλανήτη, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας απασχολούν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δώσω το λόγο στην κυρία Ουλρίκε Ρόντουστ. Την παρακαλώ να πάρει το λόγο για τρία λεπτά, βέβαια το καταλαβαίνω πως δεν είναι δυνατό, αλλά, ε, αλλά ξέρω ότι θα κάνετε την πρώτη. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ωκεανοί δεν γνωρίζουν σύνορα. Μας υποχρεώνουν να έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Μας ε, καλούν να μην ε, χτίζουμε τείχους και να απομονώμεθα. Αυτό για μένα είναι ήδη μία αξία αυτή καθευτή. Τα μέτρα για την ε, πολιτική των θαλασσών έχουν να κάνουν με την αλληλεία, με την εξόριξη βάθους και την χρήση της Αρκτικής. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία μεταξύ διαφόρων ε, δραστηριοτήτων και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ηγετικό ρόλο στη διεθνή πολιτική για τις ε, θάλασσες. Η απάντηση είναι απλή, απλούστατη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω ε, είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια δύναμη η απώλεια θαλάσσιας ε, βιοποικιλότητας και η αποδυνάμωση των οικοσυστημάτων της θάλασσας παίζει μεγάλο ρόλο στην, ε, στο κλίμα. Τις τους τελευταίους μήνες τα λίματα στη θάλασσα έχουν γίνει προτεραιότητα. Επιτέλους, σε μία ε, αποστολή διαπίστωσα ότι ένα ε, ε, ψάρι μπορεί να φά, καταπιεί πολλά ε, απορρίμματα. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να πνίγουμε τα ψάρια. Και επίσης έχουμε και τις εκπομπές από, το, από τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα βλέπω αυτά στη χώρα μου στην περιοχή μου, μπροστά στην πόρτα μου στο Σλέσφι Χολστάιν. Στα πλαίσια της παγκόσμιας, ε, της ε, γενικής ανακοίνωσης για τη διεθνή πολιτική των θαλασσών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος δεσμεύονται να δράσουν από πλευράς της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του G7 και των περιφερειακών συμβάσεων για τις ε, θαλάσσιες περιοχές. Όπω αναφέρθηκε ήδη, αυτό ο διεθνή, αυτός ο έχει κεντρική σημασία, Για το πρόβλημα είναι αναγκαστικά παγκόσμιο. Και αν δούμε και τους στόχους ανάπτυξης του, των ΟΕΕ, τις αποφάσεις του G20, του G7 και τις διάφορες άλλες ε, περιφερειακές συμφωνίες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να υπάρξει μία συνολική προσέγγιση. Αυτή την προσπάθεια πρέπει να την αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερε απαντήσει πρέπει να δώσουμε, για παράδειγμα, για την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών στη θάλασσα. Από πού όμως να ξεκινήσουμε. Πολλά έχουμε να κάνουμε και είναι πολύ μικρές οι ουσίες, ε, είναι τα μικροπλαστικά και δυστυχώς το 94% των λιμάτων καταλήγουν στη θάλασσα και στο βυθό των θαλασσών. Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί λοιπόν με απλά μέσα. Δεν είναι απλό βεβαίω. Αλλά εμείς εδώ συγκεντρωμένοι πρέπει να έχουμε ένα μόνο στόχο. Να διασφαλίσουμε το μέλλον του γαλάζιου πλανήτη μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της θάλασσας. Αλλά όχι μόνο με νέους νόμους. Έχουμε αρκετούς νέους νόμους. Πρέπει να δράσουμε με συνέπεια για να εφαρμόσουμε αυτούς τους νόμους. Να ελέγξουμε την εφαρμογή τους και ενδεχομένως να υπάρχουν και κυρώσεις και μάλιστα σοβαρές κυρώσει. Χρειαζόμαστε τις ε, θάλασσες και τους ωκεανούς για να επιβιώσουμε. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ulrike. Ευχαριστώ πολύ, Ουλρίκε. Σεβάστηκες και το χρόνο σου. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, διάφορους εμπειρογνώμονες ε, και ενδιαφερομένους ε, φορείς και θα ακολουθήσει βέβαια και μία ώρα ερωταπαντήσεων στη συνέχεια, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανταλλαγή απόψε μεταξύ ακροατηρίου και πυρογνωμόνων. Σε κάθε πυρογνώμονα θα δώσω πέντε λεπτά το πολύ. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Στίβ Τρέντα από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω ενώπιόν σας. Σας ευχαριστώ επίσης ε, που ε, διαθέτετε και χρόνο για να μας ακούσετε. Ε, θα κόψω την ομιλία μου ε, για να μην περάσω το πεντάλεπτο, άρα αφήνω τα εισαγωγικά και πηγαίνω στην ουσία. Η γαλάζια καρδιά του πλανήτη μας αντιμετωπίζει προβλήματα και για να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει να βελτιώσουμε την διαχείριση. Βλέπω τρία βασικά θέματα που θα μας επιτρέψουν να το πετύχουμε. Πρώτον, νομίζω θα ήταν ένα ασφάλμα να μην έλεγα ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσει του με τις δράσεις για το κλίμα. Θα πρέπει να βαθμίσουμε τι προσπάθειες ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην ξεπεράσει την αύξηση των δύο βαθμών ε, καλύτερα από το 1,5 βαθμό η θερμοκρασία στον πλανήτη. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση των ε, ανανάσιμων πηγών ενέργεια, σε, σε μείωση των ρεκτών για μηδενική ε, σε άνθρακα οικονομία και πρέπει να τα λάβουμε αυτά τα μέτρα παντού και στι θάλασσε και του ωκεανού. Το δεύτερο, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα για να προστατευτεί η βιοπικιλότητα στα ανοιχτά στο βάθ των ωκεανών. Έχουμε κάνει πρόταση, αλλά στα δύο τρίτα ε, των ε, ωκεανών ε, και πάνω από το 90% της εδάτενης μάζας δεν είναι ακόμα προστατευμένο. Πρέπει να προστατεύσουμε τουλάχιστον το 30% των εδάτων των ωκεανών για να μπορέσουμε και εμείς να ωφεληθούμε από τις πολλές περισσότερες που έχει να μας παράσχει και να θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη για να δείξουν ηγετική στάση και να προωθήσουν τις δράσεις και που, που σε επίπεδο ΙΕ ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο για οικολογικά αντιπροσωπευτικό δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Ε, πρόκειται για μια ευκαιρία που δεν θα δοθεί σε πολλές γενιές για τη διατήρηση, για την πραγματική βιώσιμη χρήση και την προστασία των ζωτικών πόρων για αυτή τη γενιά και τις μελλοντικέ γενιές. Επίσης, ε, απευθύνω έκκληση στο να είμαστε διαφανείς ε, για την βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης. Υπάρχουν κάποιοι που αδίστακτα κερδοσκοπούν ε, και πολλές φορές δρούν χωρίς να μπορεί κανείς να τους εντοπίσει. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε σε όλες ε, τις χώρες ε, τις αρχές που θα μπορούν να ελέγχουν για να βλέπουν ποιος, που, πώς κάνει τι. Και θέλουμε να έχουμε απλές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της διαδικασίας διαχείρισης της Έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Έχουμε παραδείγματο χάρη την ενιαία δημοσίευση ε, βασικών ε, πληροφοριών για τις άδειε αλίευσης ε, των σκαφών. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και δεν είναι και δαπανηρό, είναι δωρεάν. Επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί παγκόσμιο αρχείο μητρό των νεολογημένων σκαφών. Θα πρέπει να πάρουν δράση οι κυβερνήσει, περιφερειακοί ε, οργανώσει αλληλείας ε, και γενικώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να έχουμε ε, καταγραφή όλων των σκαφών. Και αυτό έχει πάρα πολύ μικρό κόστος, αλλά μπορεί να μεταμορφώσει την κατάσταση. Επίσης, σημαντικό είναι και σε ό,τι την εξόρυξη ε, στα νυχτά και σε όλα τα άλλα επίπεδα να ε, βοηθήσουμε ώστε να μην παρακάμπτουν με τις σημαίες ευκαιρίες ορισμένοι ε, τους κανόνες, να μην απειλείται έτσι η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια, η βιοπικιλότητα. Αυτά απαιτούν την δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα μητρώα τα, τα αναλαμβάνουν ε, την ευθύνη για τα κράτη, μάλλον αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Υπάρχουν δέσμες μέτρων που μπορούμε να εφαρμόσουμε ευθύ αμέσως και μπορούμε να είμαστε πρωταθλητέ και πρωτοπόροι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε που ιδρύθηκε άλλωστε η Ένωση, έδειξε ότι είναι μια δύναμη για το καλό. Πολλέ φορέ χρησιμοποιεί και ε, την, ε, το εμπορικό τη σήμαν, θέλετε, για να δώσει το καλό παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε δυναμική ηγεσία στο παγκόσμιο προσκήνιο, να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη αλία το κάναμε, χρειαζόμαστε αντίστοιχο όραμα και ε, πρωτοβουλία για εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας των Παρισίων για μια νέα συμφωνία των Εθνών ε, για ε, τα βαθέα ύδατα και να μην υπονομεύονται πλέον οι προσπάθειες που γίνονται από ορισμένους. Ευχαριστώ. Thank you very much, Steve. Now Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω λόγο στην πρώην Επίτροπο Μαρία Δαμανάκη που είναι επικεφαλής του οργανισμού Nature Conservancy. No. Okay. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γκάμπριελ. Είπα ότι όσο μεγαλώνω, μου είναι πολύ πιο εύκολο να μιλώ όρθια. Κύριε Επίτροπε Βέλα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητή κυρία Μάισνερ, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το κτίριο και να βλέπω να τα καταφέρνει τόσο καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ζωντανή, αλλά και δυναμική και ε, ζωντανή, ζωηρή όπως η ωκεανή. Είμαι πολύ ευτυχής και ελπίζω το ίδιο να συνεχίσει και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές. Ας το ελπίσουμε τουλάχιστον. Εδώ θα σας μιλήσω για να σας πω ότι εκπροσωπώ μια μεγάλη περιβαλλοντική οργάνωση, μία από τις μεγαλύτερες που έχει έδρα στις ΗΠΑ, τη Nature Conservancy, εκπροσωπούμε, είμαστε μάλλον παρόντες σε 72 χώρες και είμαστε μοναδικοί γι' αυτό. Από τότε που έφυγα από τις Βρυξέλλες έχω μεταβεί παντού. Αυτά που θα σας πω λοιπόν ε, είναι πράγματα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε και είμαι πολύ υπερήφανη γιατί όπου και να πήγα είδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ηγετική ε, δύναμη για την διακυβέρνηση των ωκεανών και την βιωσιμότητα των ωκεανών και ήθελα να πω ιδιαίτερα στους νέους ότι θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα μου υπενθύμησε ότι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ ε, ψηφίσαμε την ε, νέα κοινή αλλιευτική πολιτική, η οποία και ισχύει. Άρα τα καταφέρνουμε. Παρακολούθησα τους ε, νέους που μας είπαν «Κάντε κάτι». Μα κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όπως είπε και ο Επίτροπος Βέλλα, έχουμε προοδεύσει και προσβλέπουμε στο μέλλον με αισιοδοξία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και καταφέρνουμε πολλά. Χρειαζόμαστε περισσότερα φυσικά. Απειλούνται οι ωκεανοί, βεβαίως, και έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές να αντιμετωπίσουμε. Το κλίμα έχει αλλάξει άρδιν, άρα όπως είπε και ο κύριος Λέφερ, δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε σε σχέση με τον βιώσιμο αναπτυξιακό στόχο 14 αν δεν τον συνδέσουμε με άλλους ε, στόχους. Οι κλιματικές αλλαγές ισχύουν και μας ε, κατακλείζουν. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Ζουάου, χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία για να τα καταφέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ένας μείζων οργανισμός, αλλά οι ωκεανοί δεν έχουν σύνορα. Είναι μία έννοια που ξεπερνάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Νομίζω ότι εάν θέλουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον, θα ήθελα να βασιστώ σε τρεις στόχους. Μπορούμε να συνεργαστούμε επ' αυτών και είμαι σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα λάβουν υπόψη αυτή την τάση. Ένας βασικός στόχος είναι 30-30, ε, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε το 30% των ωκεανών μέχρι το 2030 και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για την βιοπικιλότητα αλλά και για την ίδια τη γαλάζια οικονομία, γιατί αν οι ωκεανοί δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η υγεία των ωκεανών έχει μεγάλη σημασία, 30% λοιπόν μέχρι το 2030. Μετά έχουμε την ε, σύμβαση, τη συνθήκη ανοιχτών θαλασσών. Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη και συνεργάζομαι και εγώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ηγετική δύναμη υπέρ της Σύμβασης Ανοιχτών Θαλασσών με βάση την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης και της βιωσιμότητας και φυσικά αποτιμώντας το τι συμβαίνει. Βεβαίως χρειαζόμαστε και χρηματοδότηση, το είπαν και οι νέοι μας. Τα χρήματα είναι κάτι το σημαντικό, το ξέρετε, αλλά για να προστατεύσουμε τους ωκεανούς υπάρχει και ένα εμπλεκόμενο κόστος. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει πια δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό θα πρέπει να μοχλεύσουμε τα χρήματα που διατίθενται για τους ωκεανούς. Ε, υπάρχει με ένα ιδιαίτερο ομόλογο το επωνομαζόμενο ε, γαλάζιο γαλάζιο ομόλογο στις Σεϊχέλες. Τώρα θα μεταβώ στο Μεξικό και θα δείξω τι γίνεται στο Κανκούν, τι γίνεται στις ε, κοραλιογενείς περιοχές και φυσικά υπάρχουν και πριμοδοτήσεις εκεί όπου χρειάζεται. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε καινοτομίες και χαίρομαι για τη Γενική Διεύθυνση ε, ΜΑΡΕ προβάλλει την καινοτομία. Πολλά αλλάζουν και χαίρομαι γι' αυτό. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον Επίτροπο Μοέδας που μίλησε για την Σίλβια Έρλ, η οποία κατοικεί στις ΗΠΑ και η οποία είπε ότι οι άνθρωποι είναι όντα, σκεπτόμενα όντα. Ο Πλάτωνας είχε πει προερχόμαστε από τη θάλασσα και θα επιστρέψουμε στη θάλασσα. Το ξέρουμε αυτό. Αποτελεί μία πραγματικότητα. Είμαστε θαλάσσια όντα λοιπόν, ας είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και ας κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε και εμείς Μαρία. Mr. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μάτινσεν από, τη από την ε, ΦΑΟ και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μάισνερ, Επιτροπή, Προηγούμε παρελθόντες και παρόντες, για να ε, παραφράσω και τα λόγια του κυρίου Φαρία. Κυρίες και κύριοι, Τέσσερα είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Εάν θέλουμε βιώσιμη διατροφή και ε, επιστημιστική ασφάλεια για όλους. Τα τέσσερα βασικά ζητήματα καταρχάς επηρεάζονται και από τέσσερις μείζονος σημασίας παράγοντες. Πρώτα απ' όλα η αύξηση του πληθυσμού και όπως όλοι ξέρουμε θα φτάσουμε τα 10 δις το 2050 το δεύτερο είναι η κλιματική αλλαγή. Όλοι καταλαβαίνουμε την ε, σημασία και τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει στους ωκεανούς και τις κοινότητές μας. Το τρίτο είναι η βιοπικιλότητα που σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το μέλλον και με τις λύσεις και το τέταρτο είναι η ρήπανση το πλέον προφανές ε, φαινόμενο είναι αυτό των πλαστικών και μετά βεβαίως έχουμε να κάνουμε και με τα απόβλητα που προέρχονται από την ξηρά. Το 10% μόνο έχει να κάνει με την δραστηριότητα των ίδιων των ωκεανών και τους ωκεανούς και με τα απορρίμματα των ε, αλληλευτικών εργαλείων ή της αλίας. Και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτά τα τέσσερα βασικά ζητήματα όλα έχουν να τέσσερις υποδιαιρέσεις κοινωνικο-οικονομικές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως σκέφτομαι τα δικαιώματα των πληθυσμών, των κοινοτήτων, τα θέματα του φύλου, της ισότητας των φύλων. Οι μισοί άνθρωποι στον κόσμο στην στον τομέα της επεξεργασίας των προϊόντων της αλίας είναι γυναίκες και η νεολαία. Η απασχόληση της νεολαίας, που είναι ένα άκρο σημαντικό ζήτημα. Κάτι λίγο πιο καθημερινό, το θέμα των ποιοτικών στατιστικών. Διότι σε αυτές βασίζουμε όλες τις αποφάσεις μας. Και το τρίτο είναι πιο ανησυχητικό είναι η επισητιστική ασφάλεια. Βλέπουμε νέα στοιχεία να αναδύονται με διαφορετικό ένδυμα κάθε φορά. Ας πούμε η αντίσταση στα αντιβιωτικά που έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις αλλά αφορά και την αλία και τους ωκεανούς προφανώς. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω το τέταρτο στοιχείο που συμπεριλαμβάνει τα τρία προηγούμενα το τεράστιο χάσμα ανάπτυξης τη διαφορά που ακόμα παραμένει μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Τα τέσσερα αυτά μείζωνο σημασία ζητήματα έχουν να κάνουν με τις θάλασσες και κυρίως την παράνομη αναρχή και μη ρυθμισμένη αλία. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο τμήμα του μεγαλύτερου πάζλ και είναι μία ανοιχτή πληγή. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και τα υπόλοιπα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειές μας. Έχουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο που ανέφερε πριν ο Στίβ. Έχουμε τις διάφορες υποσυμφωνίες που ανέφερε προηγουμένως και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προηγουμένως και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν ε, υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά τη. Αλλά και από χώρες όπως η Σουηδία ξεχωριστά. Ε, ένα μέρος της λύσης είναι οι οργανισμοί προγραμματισμού της αλίας. Εάν χρηματοδοτηθούν σωστά, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως μόνο ένα μικρό τμήμα τους χρηματοδοτείται σωστά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο θέμα είναι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που το καθορίζουν ως αρμοδιότητα και προνόμιο τα εθνικά κυρίαρχα κράτη-μέλη. Τα τελευταία 25 χρόνια επιτύχαμε πρόοδο, ιδίω στο ε, νότιο ημισφαίριο και σε ένα μέρος του βορείου, όμως στο νότιο ημισφαίριο τα πράγματα αντιστράφηκαν. Η πρόοδος οπισθοδρόμησε η αλληλευτική ένταση και δραστηριότητα προχώρησε από τα βόρεια στα νότια. Η κατάσταση των αποθεμάτων δεν βελτιώνεται. Δεν ε, τα πάει και άσχημα, αλλά δεν μπορούμε να επιζήσουμε με το 1 τρίτο των ε, αποθεμάτων να αλλιεύεται. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Εδώ γύρονται δύο ζητήματα. Οι απομακρυσμένες θάλασσες και οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Απλώς πρέπει τώρα να το εφαρμόσουμε και χρειαζόμαστε και τους απαραίτητους πόρους. Το τρίτο ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Οι παράκτιες κοινότητες, οι γαλάζιες όπως έχουν ονομαστεί, οι μικρή κλίμακας αλία, οι κοινότητες που βασίζονται στην αλία ε, κοινότητες μεταναστών, 25% ε, των ανθρώπων που ζουν από την αλληλευτική βιομηχανία βασίζονται σε αυτές τις δραστηριότητε. και τα μισά αποθέματα τα αλλιεύει ο αναπτυσσόμενος κόσμος και τα καταναλώνει ο ανεπτυγμένο. Ενώ το άλλο μίσο το αλλιεύει ο ανεπτυγμένο κόσμος και εκεί έχουμε 95% του πληθυσμού. Είναι περίπλοκο αυτό το ζήτημα και αυτή η ισορροπία εδώ. Χρειαζόμαστε νέε λύσει και εργαζόμαστε σκληρά για να το πετύχουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε υποστήριξη υποστήριξη από οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει με την αυξημένη ε, προσφορά ε, των προϊόντων στο μέλλον, κυρίω από την πηγή τη υδατοκαλλιέργεια. Χρειαζόμαστε πιο πολλά ψάρια για τον πληθυσμό που αυξάνεται. Δεν θα τα ε, πάρουμε από την αλεία στι θάλασσε και του ωκεανού, θα προέλθουν από την υδατοκαλλιέργεια. Ε, εδώ και την υδατοκαλλιέργεια. Εδώ υπάρχει θέμα οικολογικού αποτυπώματο των παραγωγικών συστημάτων τη υδατοκαλλιέργεια. Εάν όμω το βάλουμε στόχο, μπορούμε να σχεδιάσουμε τέτοια παραγωγικά συστήματα που δεν θα βαραίνουν τόσο πολύ το περιβάλλον. Το αποτύπωμά τους θα είναι ε, καλύτερο από ό,τι σήμερα. Και θα έχουμε βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων και στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο κ. Πασκουάλ Γόναντεφέο, Διευθύνων Σύμβουλος της Κονατέκο ΕΣΠΕ. Για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πω ότι είναι ε, για μένα πραγματικό προνόμιο να βρίσκουμε εδώ. Είμαι πρόεδρος ενός τερμινάλ του Μιλάνου του λιμένα της Νάπλης που ανήκει σε μια πολυεθνική εταιρεία που εξυπηρετεί το εμπόριο και συνδέει χώρες από όλο τον κόσμο. Επίσης είμαι πρόεδρος ε, της περιοχής της ε, Καμπανίας. Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι επιχειρήσεις ε, της επιμελητίας και συνδέουν τους λιμένες με τις οδικές μεταφορές και σε μία από τις πιο σημαντικές ενώσεις της Ιταλίας που εδώ και πολύ καιρό ασχολείται για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Σήμερα υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη σχετικότητα ε, για την θαλάσσια οικονομία, το, η έννοια της γαλάζιας οικονομίας ε, που αρχίζει να αναδύεται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ε, χάρη στην μεταποίηση των ουσιών που γίνονται εμπορεύματα. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με άλλους παγκόσμιους οργανισμούς εργάζονται για να ρυθμίσουν μία σειρά δράσεων που να καθιστούν το κλάδο μας πιο βιώσιμο. Έτσι λοιπόν ε, είναι γνωστή η στόχη. Το 2020 προβλέπεται μείωση του ποσοστού ε, του θείου ε, από το 3,5% στο 0,5%. Όμως δυστυχώς πρέπει να αναφέρω ότι στο παρελθόν οι πολιτικές των κυβερνήσεων ε, συχνά δεν επένδυσαν σε υποδομές που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μεταφορών μέσω της θάλασσας ε, που ρηπαίνει περισσότερο, υποστηρίζοντας αντίθετα τρόπους μεταφοράς ε, χερσαίους με κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος για τις μελλοντικές γενιές σήμερα η συνειδητοποίηση της σημασίας μιας ε, αηφόρου ανάπτυξης των λιμένων ε, και για τον θελέσιο μεταφορών ε, αναδύεται λένε και περισσότερο. αποτελούν παράδειγμα των πολιτικών των ναυτιλιακών εταιριών που στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε αυτές οι πολιτικές έχουν να κάνουν με τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και στη δραστική μείωση των αποβλήτων ε, που οδηγούνται στα λιμάνια. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα της εταιρεία του μήλου όπου συμμετέχω. Έχουμε ε, μια εταιρεία που ανήκει στην MSC. Έχουμε εγκαταστήσει μηχανές για να ε, υπάρξει αναγέννηση βιώσιμη και οικονομική ε, των αποβλήτων που παράγονται επί του σκάφους και είναι δυνατόν να μειώσουμε ε, τον όγκο μέχρι τον 90%. Και αυτά χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ε, και πάρα πολλά τερματικά στους λιμένες έχουν στρέψει τις πολιτικές τους προς την απόκτηση μέσων να τροφοδοτούνται δηλαδή τα πλοία με ηλεκτρισμό, ηλεκτρικό ρεύμα και αντικαθιστούν τα παραδοσιακά καύσιμα. Επίσης εφαρμόζουν τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον έλεγχο των μηχανών. Σε αυτή την οπτική, οι εθνικές και κοινοτικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν ε, με τις governance των λιμένων, ε, προκειμένου να παρέχονται περισσότερες κατάλληλες υπηρεσίες και ενεργειακά αποδοτικές που ε, να βοηθούν τις, ευκαι... τις οι πολιτικές των ε, θεσμικών οργάνων θα έπρεπε λοιπόν ε, να ακολουθούν δύο άξονες. Την υλοποίηση δημοσίων υποδομών, ε, δηλαδή εξοπλισμό για ε, ηλεκτρικό ρεύμα και ε, να υπάρχουν ε, αποθήκευση φυσικού αερίου, πολυτροπικές διασυνδέσεις με την επικράτεια, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία και με κάποια καθυστέρηση έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί για να δημιουργηθούν αυτές οι αποθήκες για το ευρωπημένο φυσικό αέριο. Και από την σκοπιά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι οικονομικοί φορείς που ε, ασχολούνται μόνο με την ναυσιπλοεία, με τις θαλάσσιες μεταφορές, ε, να κάνουν αξιοσημείωτες επενδύσεις, δηλαδή ε, να δοθούν και κίνητρα σε αυτούς τους επιχειρηματικούς φορείς να επενδύσουν σε τεχνολογικές λύσεις που να μπνέονται από τη γαλάζια οικονομία. Λέγεται ότι η γαλάζια οικονομία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένως, η αναγκαιότητα υπάρχει για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά όλοι μαζί. Όμως ε, υπάρχει και υποχρέωση, λαμβάνοντα ε, υπόψη την ιστορική στιγμή που θα βιώσει η χώρα μου αυτή την εβδομάδα, ε, να προσέξουμε τι προσφέρεται από την Κίνα, η λεγόμενη πρωτοβουλία Bent Elrod η Κίνα και θέλω να το επενθυμίσω την προηγούμενη δεκαετία παρουσιάστηκε σε όλο τον κόσμο στο παγκόσμιο εργοστάσιο με χαμηλό κόστος εργασίας και ε, ποιότητα παραγωγής. Έτσι λοιπόν μπόρεσε να αγοράσει τις τεχνολογίες δυτικών εταιριών. Και αφού κατέκτησε την τεχνολογία, προέβησε αναβάθμιση στην αλυσίδα αξίας και στην ποιότητα των προϊόντων και παρουσίασε στον κόσμο νέε τεχνολογίες πιο πολύπλοκε από τις δυτικέ. Το 2014 ξεκίνησε ένα τεράστιο φαρανικό σχέδιο ε, χρησιμοποιώντας 120 ε, δισεκατομμύρια στι στις αγορέ, ε, και αυτή τη στιγμή μόνο 70 χώρες, αλλά σκοπεύει να συνάψει 100, συμφωνίες με 120 χώρες για να δημιουργήσει το Silk Road, αλλά και το One Belt, One Road, για να, συνδεθεί, να με την αγορά της. Ε, βλέπουμε ότι η παρουσία στο εσωτερικό της Ένωσης των κρατών που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Κίνα, πέρα από το ότι θα υπάρξουν μειονεκτήματα και απώλεια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές μπορεί και να αποδυναμώσει πολύ τη δράση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας. Και δεν είναι τυχαία και η προσοχή που δίνεται στην Ελλάδα ε, δυστυχώς έχει παραχωρήσει ένα στρατηγικό λιμένα στην Κίνα, τον Πειραιά και δυστυχώς ε, υπάρχει και επιρροή και στις πολιτικές αποφάσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιε ε, χώρε ε, που στην αρχή, κάποιες χώρες που έχουν δείξει θυσιασμό, όπω το Πακιστάν, Σιέρα Λεόνε, το Μπαγκλαντές ε, και άλλες, στη συνέχεια κύρωσαν τις δεσμεύσει τους, επειδή αυτά, αυτά τα προγράμματα, τα σχέδια των υποδομών θα χρεώναν υπερβολικά τι χώρε. Σήμερα μιλάμε στην Ιταλία και για την ανάλυση ωφέλους. Αφού έκαναν τέτοιες αναλύσεις, γύρισαν την πλάτη στην οδό του μεταξιού. Εγώ, όντα Ευρωπαϊστή, εύχομαι η Ευρώπη να παραμένει πάντοτε πιο ενωμένη για να έχει την ικανότητα και την πολιτική βούληση να υλοποιήσει όλε τι απαραίτητε δράσει και να δώσει του αποφασιστικού αγώνε για να κερδίσει την, αυτήν τη γαλάζια οικονομία. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους ε, ομιλητές. Αρχίζει αμέσως η συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις. Άμε χάλια από χρόνο που δείχνει ότι δεν είμαι καλός πρόεδρος γιατί δεν σας διέκοψα. Θα προσπαθήσουμε στο γύρο των ερωταπαντήσεων να κερδίσουμε χρόνο. Παρακαλώ ποιος θέλει το λόγο να σηκώνει το χέρι του και να περιμένει να του δίνεται ο λόγος. Σας παρακαλώ να κάνετε ερωτήσεις πάρα πολύ σύντομες και όχι μεγάλες τοποθετήσεις ε, για το τι πρέπει να γίνει. Συγκεκριμένες ερωτήσεις να συστήθετε πρώτα και να μας πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας κάθε φορά. Ο Τζουζέπε Σκινότη από την Nova Meet, παρακαλώ. Thank you, Chair, and good afternoon to the, all attendees, especially... Ευχαριστώ και καλωσορίζω και όλους τους προσκεκλημένους και όσους ήρθαν, κυρίως τους νέους. Πολύ γρήγορα, είμαι ο κύριος Σόντι, πρώην μηχανικός και εργάζομαι για Nova Novamit. Και ασχοληθήκαμε με τις εναλλακτικέ προϊόντων ψαριών και κρέατος που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Μας ενδιαφέρει στην Ευρώπη να δούμε πώς ε, έχει αυξηθεί στη διατροφή μας κατανάλωση προϊόντων κρέατος και ψαριού. Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Οργανικού Υγείας δείχνουν ότι είναι, δείχνουν ότι είναι ανησυχητικά ε, όσα συμβαίνουν για όλους μας και ότι είμαστε στην, στην κακό δρόμο για να προστατεύσουμε τους ωκεανούς. Υπεραλίευση, απώλεια της βιοπικιλότητας, ε, ρήπανση από τα μικροπλαστικά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ωκεανοί υπάρχουν εδώ και δύο εκατομμύρια χρόνια, ενώ η ανθρωπότητα ενώ και δύο εκατομμύρια μόλι χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν το 2019 πρέπει κάτι να αρχίσει να κάνει για αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Έχουμε και ε, δυνατότητε και ευθύνε. Είναι και τύχη που θα μπορούσαμε ε, να μείνουμε στην ιστορία ω η πρώτη γενιά ανθρώπων που αντέστρεψαν την τάση των αλλαγών του κλίματο για τα παιδιά μα και το μέλλον και προτού ε, γίνουμε 10 δι άνθρωποι στον πλανήτη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει νέε ευρωπαϊκές τεχνολογικέ λύσει για να χειριστεί καλύτερα του πόρου των ωκεανών μα. Στην Ευρώπη έχουμε ταλέντο, δημιουργικότητα και τη δύναμη για να φέρουμε αυτέ τι λύσει στην αγορά και να σώσουμε του ωκεανού μα. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερο, η καλύτερη κινητήρια δύναμη για να σώσει τους ωκεανούς μας. Ε, παρά τη μεγάλη κρίση τη ανθρωπότητα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ομαδοποιήσουμε λίγο τις ερωτήσεις ανά για να δοθούν απαντήσει. Το έδρανο 115. Επειδή δεν ξέρω τα ονόματά σα, θα λέω το αριθμό του εδράνου στο οποίο κάθεστε. Εξαιρετική η διάσκεψη. Υπάρχει ένα ταμπού. Το οξυγόνο δεν το συζητάμε το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, συζητάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ζωή το οξυγόνο. Η θάλασσα μας δίνει το οξυγόνο. Μήπως θα πρέπει να αρχίσει μια πολύ μεγάλη έρευνα για το οξυγόνο και μάλιστα την παραγωγή οξυγόνου από τους ωκεανούς. Ευχαριστώ. 248. Pierre Dumoulin, je εκπροσωπώ μια ε, τοπική ε, ε, επιτροπή στις Βρυξέλλες γιατί δεν μιλάμε για όλα τα πυρομαχικά. 35.000 ε, ετών στα ανοιχτά του ΚΝΟΚ ε, ανάμεσα στην ε, Σκοτία και την Ιρλανδία και στη Βαλτική. Έχουμε δανούς ψαράδες, τραυματίες και πάρα πολλά επεισόδια. Οι δανοί ψαράδες υφίσταται πολλές μεγάλες δηλητηριάσεις και έχουν πρώτες βοήθειες κατά των δηλητηριάσεων ε, τύπου υπερίτη ε, στα σκάφη τους, στα λεφτικά. Η Φιλανδία ήδη δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οβίδες έχει βγάλει ε, από εκεί που περνάει το, ο αγωγός Nord Stream 2 στα χωρικά της Ήδατα. και αλλού. Είναι πολλά τα τοξικά πυρομαχικά στην Αδριατική, στην Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή οι Άπωνες είναι οι μόνοι ε, που ανακτούν ε, αυτά τα πυρομαχικά για να τα καταστρέψουν ε, από τα βάθη των ωκεανών. Δεν θα μιλήσω για τις λίμνες της Ελβετίας ή για την Αμερική. Αυτά θα τα αναλάβει ο κύριος Τραμπ. Θα πρέπει η Ευρώπη επιγόντως να βιαστεί, αν δεν θέλουμε να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, να βιαστεί τι εννοώ στο Οικαιογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας έχει γίνει μια έρευνα που λέει αν, βγει το 1 έκτο, το αν δεν βγει το 16% ε, θα πεθάνει για 30 χρόνια η Βαλτική αν αδρανίσουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιληφθεί. Ε, με ρομπότ θα μπορούσε να γίνει αυτό, οι Κινέζοι ενδεχομένως, μια Αμερικανική εταιρεία, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Θα απαντήσουμε στις τρει αυτέ ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ ερωτήσεις να κάνετε, όχι τοποθέτηση και εξήγηση 1,5 λεπτό, γιατί δεν θα προλάβουμε να ε, ακούσουμε τις απαντήσεις. Ποιο θέλει να απαντήσει. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Γκαμπριέλ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Ήδη εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ορίζοντα 2020, ε, λέει ο Ζωάγκυρα Ματσάδο, για την έρευνα στους ωκεανούς. Και αυτά που σας είπα, ε, το ακούσαμε και στην εισαγωγή από τον Επίτροπο, τον κύριο Μοέδας. Στο νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπης, όπου αυξάνεται, σύμφωνα με τις πρότασεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο προπολογισμό, έχουμε αυτό τον ειδικό στόχο ε, για τους ωκεανούς. Να έχουμε αυτή την έρευνα χάρη στην πολιτική ηγεσία των ε, Επιτρόπων Βέλα και Μοάδας, σε αγαστή συνεργασία. Και ο συνάδελφος Ζάιρικ Πακέ είναι στο επόμενο πάνελ και θα μπορέσει σίγουρα να σας πει περισσότερα. Αυτή είναι όμως η πρώτη φορά όπου θα έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα αναγνωρισμένο παγκοσμίω ως από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα και θα έχουμε ειδικέ αποστολές αυτή τη φορά για τους ωκεανούς. Ευχαριστώ. Άλλος. Ε, Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο που μίλησε προηγουμένως και να πω για τις τοξικές ουσίες και για τα πυρομαχικά κατάλοιπα. Υπάρχουν χειρότερα προβλήματα στους ωκεανούς. Υπάρχουν τα πυρηνικά απόβλητα, λόγω χάρη. Ξέρετε ότι στη δική μου τη χώρα, την Πορτογαλία, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ε, ολόκληρες δεξαμενές με τοξικά απόβλητα από πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτά καλά θα, θα τα συζητήσουμε. Το έχω ξαναπεί στο Κοινοβούλιο. Το έχω πει. Δεν είναι μόνο τα τοξικά πυρομαχικά απόβλητα που ή μπορεί να είναι ανώδυνα. Ε, εδώ και στις ευρωπαϊκές ακτές έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως τα μπιτόνια που σας είπα που ανακαλύπτουμε. Και καλό θα ήταν να το δούμε εν και της ερχόμενης εβδομάδας. Άλλα σχόλια, κυρία Δαμανάκη. I would like just to Θα ήθελα απλώς να πω ότι έχει δίκιο ο κύριος εκεί. Δεν έχουμε αρκετά επιστημονικά στοιχεία ούτε αξιολογήσεις που μπορεί να συνδέουν ε, την κλιματική αλλαγή με τα μεγάλα βάθη των ωκεανών. Έχουμε μελετήσει τις παράκτης περιοχές, ε, τα ε, κοραλιογενή νησιά και άλλους βάλτους θάλασσες κοντά στη θάλασσα, αλλά για τα μεγάλα βάθη των ωκεανών δεν έχουμε μελετήσει την κλιματική αλλαγή. Αν υπάρξουν επιστημονικά στοιχεία, σίγουρα θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Και τα πανεπιστήμια μπορούν να βοηθήσουν και τα Ινστιτούτα και συμφωνώ με το ΖΟΑΟ. Ο κύριος Μάτο. η κυρία Ουρίκε Ρόντος. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τα τοξικά ε, πυρομαχικά και τις τοξικές ουσίες. Ε, εγώ είμαι από το Σλέσφικ Χολστάιν ε, που βρέχεται από τη Βαλτική. Και στη δική μου περιφερειακή πολιτική, στην Περιφερειακή Βουλή, συζητούμε και με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κρατηδίου από τότε που ασχολούμαι με την πολιτική. Και βλέπετε από τα γκρίζα μου μαλλιά ότι είναι πολλά τα χρόνια. Έχω μάθει λοιπόν πάντα ότι το ταμείο είναι μείον. Ό,τι και να θέλεις, ό,τι, όσο και μεγάλο να είναι το πρόβλημα, ε, ο ένας ε, το παραπέμπει στον άλλον και ε, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε χρήματα. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που ακούω διαμαρτυρίες και δυνατές φωνές που διατρανώνουν θα πρέπει να πιάνουν περισσότερο τόπο τα χρήματά Μα Συμφωνώ απολύτως. Επιγόντως θα πρέπει να δράσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε νόμους λογικούς για την αλία ότι και δεν μπορούν μετά να ψαρεύουν οι αλίες επειδή είναι καταδηλητηριασμένα τα ψάρια. Ε, Δυστυχώ δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για ερωταπαντήσει, γιατί μιλήσαμε εμεί πολύ. Θα πρέπει να δώσουμε τώρα το λόγο στο δεύτερο πάνελ για τις ε, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ από το πρώτο πάνελ.